Um, θα ξεκινήσουμε. Πάλι έχουμε το web stream, την μετάδοση από το διαδίκτυο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Δεν είμαστε και τόσο πολλοί, αλλά ελπίζω ότι θα έρθουν και άλλοι σε το χρόνο. Το θέμα μας είναι πλατφόρμα δημοσίου συμφέροντος οδηγία οικουμενικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα εργασίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, της ΕΝΙΣΑ. Καλώς ορίζω θερμά τον κύριο Ούντο Χέλμπρεχτ, το διευθυντή της υπηρεσίας, ο οποίος ήρθε αεροπορικός. Ξέρετε πόσο χρόνο αφιερώνουμε στη συζήτηση για την υπηρεσία σας εδώ στο Κοινοβούλιο για θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών που τους δίνουμε μεγάλη, μεγάλη σημασία σε μια διαρκώς μεταλλασσόμενη κατάσταση. Και έχουμε ενημερώσει, Ανδρέας, και την ε, ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου ότι είναι ένα θέμα στο οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία. Και ότι πρέπει να κοιτάξουν ε, σε όλους τους τομείς τριμερούς διαλόγου αυτή τη διάσταση. Η γραμματεία μας έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο ενημερωτικό, να το δείτε και μια και μεταδίδεται δι- του διαδικτύου η συνεδρίασή μας. Το δείχνω στις κάμερες. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν ως έγγραφο ενημερωτικό. Ούντο, θες να μας, να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες και μετά θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για την ε, εισαγωγή αυτή, Πρόεδρε. Σήμερα θα σας ε, μιλήσω για ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς της ΕΝΙΣΑ. Θα σας εξηγήσω το εξής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κανονισμός προστασίας των δεδομένων ε, και η οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών συζητώνται αυτή τη στιγμή ε, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Αυτά τα θέματα σχετίζονται με τις δραστηριότητες μας. Ας δούμε το πιο ευρύ πλαίσιο. Ε, έχουμε την στρατηγική ασφάλεια των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την προσέγγιση της νέας ψηφιακής αγοράς Έχουμε πολλά πράγματα δηλαδή τα οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ε, η ασφάλεια της τεχνολογίας των πληροφοριών ε, είναι το θέμα το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει και ως ενίσα, αλλά ταυτόχρονα ε, και τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσει και τους ίδιους πολίτες. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζουν την δουλειά μας, τα καθήκοντά μας, αλλά θα ήθελα να σας πω το εξής. Έχουμε τρεις στοιχεία στη δουλειά μας. Πρώτον, αναλαμβάνουμε, αναπτύσσουμε ε, project ε, τα 25-30 κάθε χρόνο, ε, τα οποία σχετίζονται με θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών και δημοσιεύουμε τα πορίσματά μας. Το δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο, δυνάμει το άρθρο 14, τα κράτη-μέλη μας ε, ζητούν με σεμινάρια ε, επιμορφωτικά, ασφάλειας ε, κλπ. Και ταυτόχρονα υποστηρίζουμε και την ομοθετική διαδικασία. και όχι μόνο την καθαρά την καθαρή διαδικασία ε, του νομοθετικού έργου αλλά και, το στάδιο της ε, εφαρμογής. Βοηθούμε για παράδειγμα σε οποιαδήποτε διαδικασία ε, παράβα, επεπαραβάση, χρειάζεται να ξεκινήσει κλπ. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Στις ε, κυβερνήσεις υπάρχουν, οι κυβερνήσεις έχουν εσωτερικές δομές, έχουμε ε, συνδέσμους, έχουμε υπουργεία, έχουμε γραμματείες κλπ. Και σε κάθε επίπεδο ξέρουμε με ποιον θα μιλήσουμε. Όμως, ε, στις επιχειρήσεις έχουμε λόμπι, έχουμε συνδέσμους, ενώσεις ε, κλπ. Αλλά εκεί δεν έχουμε μια εσωτερική δομή όπως αυτή των κυβερνήσεων. Εκεί έχουμε διάφορους ε, εμπλεκόμενους ε, με τους οποίους έχουμε θέμα να δούμε ποιος τους εκπροσωπεί. Και με τους πολίτες είναι ακόμα και δυσκολότερα τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο εδώ και δύο χρόνια έχουμε ξεκινήσουμε τον Ευρωπαϊκό Μήνα Ασφάλειας των Εξυπηρετητών, των Servers, ε, κατά τη διάρκεια του οποίου μήνα μαζί με οργανώσεις των κρατών μελών, υποστήριξη των κυβερνήσεων με την Κομισιόν κλπ. προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες. Το 2012, το 2013, 2014 και το 2015 ε, έχουμε ε, ε, συμμετοχή όλων των κρατών μελών μαζί με την Ορβηγία και την Ελβετία Οπότε προσπαθούμε ε, να διοργανώσουμε εκδηλώσεις, για παράδειγμα τον Οκτώβριο, ε, πολλά κρατημέλη, πολλοί πολίτες θα, ε, κάθε Οκτώβριο τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν έτσι ώστε η πληροφορία να φτάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη και στους πολίτες μέσω των οργανώσεών τους αυτή τη στιγμή εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους που θα οργανώσουν τα επόμενα, εκδηλώσει εκδηλώσεις στα κράτη-μέλη. Οι επόμενε εκδηλώσει αυτές θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο. Ε, ετοιμάζουμε ερωτηματολόγια σε διάφορε γλώσσε. Έχουμε ήδη στις 24 ε, γλώσσες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ο δημόσιος τομέας, οι ερευνητές, ακαδημαϊκοί, συμμετέχουν, παίρνουμε τη γνώμη ε, των ε, ενδιαφερομένων και έχουμε ένα πολύ ε, και έχουμε πολύ περιεχόμενο το οποίο έχουμε να μοιραστούμε με το κοινό μας. Συμμετέχουν μη κυβερνητικέ οργανώσει, η βιομηχανία, οι πολίτε, η κοινωνία των πολιτών, κυβερνήσεις κλπ. Ο μέσο χρήστη τελικά. Ποιος είναι ο μέσο χρήστης έχουμε τέσσερις βασικές ομάδες μέσων χρηστών. Πρώτον, οι νέοι, ακόμα και τρίχρονα, τετράχρονα παιδιά παίζουν πια σε ταμπλέτες πριν καν αρχίσουν να διαβάζουν και να γράφουν, διάβασα κάπου. Ε, μετά ε, έχουμε, μάλλον έχουμε λοιπόν νέους, ε, κυρίως μεταξύ ηλικιών 10 και 20 ετών, που δεν σκέφτονται και πολύ την ασφάλεια, και αν δούμε λίγο πιο βαθιά σε αυτήν την ομάδα, γνωρίζουν από τεχνικής πλευράς τους κινδύνους, ε, ε, σκουλίκια, ιούς, ε, ε, ιδιωτικότητα κλπ. Όλα αυτά τα ξέρουν, αλλά θεωρούν ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Και είναι δύσκολο να πείσει ένα 15χρονο ε, τι συνέπειες θα έχει χρήση ε, των δικτύων 10-15 χρόνια μετά την άλλη μεριά, ε, τις προάλλες ε, έμαθα ότι το 60% των μεγαλύτερων ε, ηλικιών χρησιμοποιούν προστασία, ε, τείχους προστασίας, αντιϊκά κλπ. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχει το 1 τρίτο, έτσι, το υπόλοιπο 40% που δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους προστασία. Ε, και ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, τους γυρεότερους και τους πιο νέους, έχουμε άλλες δύο ομάδες. Έχουμε μια ομάδα ε, πολύ μορφωμένων ανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα σε καθημερινή βάση. Και από την άλλη μεριά έχουμε ένα μέσο χρήστη που χρησιμοποιούν ε, τα πολύ βασικά πράγματα, ε, συναλλαγές, τραπεζικές ε, συναλλαγές, ενημέρωση κλπ. διαφέρουν λίγο αυτές οι ομάδες μεταξύ τους. Τώρα πώς θα φτάσουμε σε αυτούς, έτσι έχουμε τέσσερις ομάδες τις οποίες πρέπει να αγγίξουμε. Ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη έχουμε ήδη εργαλεία στη γλώσσα τους ε, που απευθύνονται σε κάθε ομάδα χωριστά. Τι θα κάνουμε φέτος. Ε, έχουμε το πόρταλ με τα εργαλεία ιδιωτικότητας το οποίο συνδέεται και με τον, την εφαρμή του κανονισμού προστασίας δεδομένων. Επίσης θέλουμε να δούμε πώς οι πλατφόρμες, οι online ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να επιμορφώνουμε το κοινό, για να τους βοηθάμε και να τους ενημερώνουμε. Αυτά ως γενική εισαγωγή, μπορούμε να πούμε σε λεπτομέρειες αργότερα. Πάντως ε, το βασικό είναι ότι προσπαθούμε να συνεργαστούμε ε, και να φέρουμε σε επαφή το ευρωπαϊκό επίπεδο με τις κυβερνήσεις και τους ε, πολίτες, επιχειρήσει και, και τους, ε, τις οργανώσεις τους. Μιλούμε για εκπαίδευση. Ε, προσπαθούμε να βρούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι στο κάθε κράτος μέλος για την εκπαίδευση, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις, δράσεις, ε, τις δράσεις. Ε, από την άλλη μεριά έχουμε την διαδικασία ψηφιακή ενιαίας αγοράς. Τι σημαίνει αυτή προσπαθούμε για τους πολίτες και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την βελτίωση της συνειδητοποίησης, της ευαισθητοποίησης του κοινού και τέλος πώς μπορούμε να ε, πλησιάσουμε συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού εστιασμένα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο. Έχουμε πολλές πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη και έχουμε 510 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη. Και αν δείτε τις πρωτοβουλίες Ε, στην πρωτοβουλία που ξεκίνησαμε πέρσι έχουμε μόνο χίλια hits στη σελίδα μας. Πολύ λίγο δηλαδή. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Επίτροπος Κρούς. Ε, βλέπετε ότι είναι πολύ μικρή απήχηση. Ακόμα και οι ε, πρωτοβουλίε που λαμβάνονται στα σχολεία είναι περιορισμένου ελληνικού. Χρειάζεται να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα πολύ πιο ευρύ φάσμα του πληθυσμού. υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν κλικ στο site μας ε, κάθε μέρα για να διαβάσουν προφορίες μας, οπότε πρέπει και εμείς να φτάσουμε σε αυτούς με άλλο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλωσορίζω και τους επισκέπτες ε, από το House of Commons, από το Westminster. Καλώς ορίσατε βρισκέστε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και συζητάμε με τον Διευθυντή της ΕΝΙΣΑ σχετικά με το έργο τους και στα 28 κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη των δυνατοτήτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Και τώρα εξετάζουμε τα δίκτυα και την ασφάλεια στο διαδίκτυο του ε, εισηγητή ΣΒΑΜΠΑ. Τώρα αναμένουμε τις ερωτήσεις. Αντρέα, θέλετε να ξεκινήσετε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ καταρχάς τον κύριο Χέλπρεχτ για την εξαιρετική εισήγηση που δείχνει ότι μια υπηρεσία όπως η ΕΝΙΣΑ είναι πολύ σημαντική και για την κλασική αλλά ιδιαίτερα για την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Είναι, έχει μια πολύ ε, σημαντική οριζόντια εγκάρσια λειτουργία. Σε παρακαλώ, Ανδρέας, ένα λεπτό. Όποιος θέλει να ακούσει στα αγγλικά πρέπει να πατήσει το κανάλι νούμερο 2. Άλλες γλώσσες θα βρείτε στα διαφορετικά νούμερα από τις καμπίνες. Για να επιλέξετε τη γλώσσα σας. Θα συνεχίσω όμως στα γερμανικά, λέει ο κύριος Φαπ. Ναι, και εγώ θα ακούω στα ισπανικά του, λέει ο πρόεδρος. Ε, διαδραματίζει λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο και αξιόλογο ρόλο η ΕΝΙΣΑ, ιδιαίτερα για την ε, ψηφιακή πτυχή της εσωτερικής αγοράς. Και γι' αυτό κυρία Χέλμπρεχτ θα ήθελα να διατυπώσω δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις καταρχήν. Στο πλαίσιο, στο πλαίσιο της Οικουμενικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Δημοσίου Συμφέροντος, εσείς μπορείτε να αποτελέσετε μια πλατφόρμα ω ε, συνδετικό κρίκο δηλαδή, μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων των σχετικών υπηρεσιών. Στο επόμενο που μας διέθεσε η Γραμματεία για να προετοιμαστούμε, μας αναφέρεται ότι έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη μέσω της ΕΝΗΣΑ να κοινοποιούν στον τελικό χρήστη ορισμένα πράγματα, τα οποία όμως δεν αξιοποιούνται. Θέλετε να μας εξηγήσετε ακριβώς ποιο είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά τη γνώμη σας, δεν έχουν αξιοποιήσει τα κράτη-μέλη αυτή τη δυνατότητα. Και δεύτερον, τους τελευταίους μήνες συζητήσαμε πανελειμμένο στο ρόλο της ΕΝΙΣΑ και επί τη ευκαιρία της οδηγίας για την ασφάλεια. Η ΕΝΙΣΑ, εάν δει το φως της σήμερα σε αυτή η οδηγία και παραμένουμε αισιόδοξοι προς αυτό, θα έχει σημαντικό καθήκον για τον προσδορισμό των προδιαγραφών, των προτύπων που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλίσουν την ε, ανθεκτικότητα ή τη δυνατότητα άμυνας στην κυβερνοεπίθεση και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα πώς νομίζετε ότι μπορεί αυτή, αυτά τα πρότυπα να διαμορφωθούν κάποια στιγμή. Θεωρείτε δηλαδή ότι τα δεδομένα τα οποία αφορούν κρίσιμες ψηφιακού χαρακτήρα ε, δομές των επιχειρήσεων και ε, αποθηκεύονται, μπορούν να αποθηκεύονται ενδεχομένως σε έναν ευρωπαϊκό σερβερ εξυπηρετητή. Γιατί έχουμε τώρα μια σειρά από δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο με τρόπο κάπως συγκεχημένο η αμερικανική πλευρά. Ξέρουμε ότι αποθηκεύει πάρα πολλά πράγματα στους δικούς της ε, εξυπηρετητές. Θεωρείται ότι και η ευρωπαϊκή πλευρά μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε μία λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες της ε, ε, ανθεκτικότητας σε επιθέσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τα μέλη τα οποία θα ήθελαν να μιλήσουν μπορούν να το επισημάνουν για να φτιάξω τον κατάλογο. Εύλην και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και για την ενημέρωση που μας προσφέρατε. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές ε, προϋποθέσεις ασφαλείας και απαιτήσει ασφαλείας και όσον αφορά τη ε, διάσταση του κυβερνοχώρου αλλά και την προσφατασία των ατόμων. Διαπιστώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα και επιχειρήσεων, δεδομένα επιχειρήσεων μπορεί να είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, όλο και περισσότερο εκτεθειμένα σε επιθέσεις Και άρα τίθεται το ερώτημα με ποιον τρόπο μπορούμε να μεριμνήσουμε για την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος στην ε, διαβίβαση πληροφοριών, για την παροχή πληροφοριών των ε, πολιτών μας, πώς θα μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα τους τρόπους άμυνας και προστασίας. Αναφερθήκατε βέβαια και εσείς στο ότι πολλοί είναι οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ακριβώς συνειδητοποιήσει το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Επί παραδείγματι να αλλάζουν ε, από καιρού εις καιρών το password, τον κωδικό πρόσβασης ή ότι θα μπορούσαν να ε, εγκαταστήσουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή ένα firewall, ένα τείχος προστασίας. Πώς μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν αυτό για τον πολίτη η πληροφόρηση και πάνω απ' όλα η συνειδητοποίηση του ότι πρόκειται για κάτι το σοβαρό και το σημαντικό. Κυρία Γκραπίνη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαι εδώ ανάμεσά σας. Θα ήθελα να επιστρέψω στη Ρουμανία λέγοντας τους ε, αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε για ενημέρωση των πολιτών μας και ελπίζω να μπορέσετε να μου το πείτε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εδώ έχω μια ιδιαίτερη προσκεκλημένη, μια φοιτήτρια από το Πανεπιστημιακό Κέντρο του ΙΑΣ, του Ιασίου και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορεί να παραστήσει αυτήν εδώ τη συζήτηση. Μερικές ερωτήσεις από μέρους μου. Κύριε Διευθυντά, ε, Αναφερθήκατε σε αυτές τις διάφορες κατηγορίες ατόμων, νέους, ε, ε, ηλικιωμένους, συνταξιούχους. Ε, είπατε ότι ορισμένοι φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες πληροφορικής. Άλλοι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σε θέματα ασφαλείας στον κόσμο της πληροφορικής. Σε γενικές γραμμές ένας άνθρωπος φοβάται μπροστά στο άγνωστο. Το άγνωστο είναι αυτό που δημιουργεί φόβο. Εγώ προσωπικά έχω τρεις ερωτήσεις ε, σε αυτό το πλαίσιο. Όσον αφορά το σύστημα εκπαίδευση σε όλα τα κράτη-μέλη, δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να ενισχύσουμε τα μαθήματα πληροφορικής ε, και να διδάσκουμε όχι μόνο τον τρόπο χρήσης ε, των υπολογιστών αλλά να μαθαίνουμε στους ανθρώπους και τους κινδύνους, στην ασφάλεια, Δηλαδή να μην περιοριζόμαστε στην απλή χρήση μιας ταμπλέτας για παιδιά ηλικίας τριών ετών. Θέλω να μου πείτε και εσείς τι πιστεύετε. Δεν θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να εμβαθύνουν ε, τα μαθήματα πληροφορικής στα σχολεία ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν από την πρώτη μέρα που χειρίζονται μια ταμπλέτα ε, και τα λοιπά προβλήματα πέρα της χρήσης λοιπόν ε, να μαθαίνουν και την ασφάλεια. Δεύτερον, ε, οι κυβερνήσεις ε, δεν θα πρέπει να δείξουν κάποιο ενδιαφέρον στο να δημοσιοποιήσουν αυτές τις ε, πληροφορίες τους πολίτες τους γιατί σε τελική ανάλυση κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση θα έπρεπε να ενημερώνει τους πολίτες της. Και τελευταία ερώτηση τρίτον, Έχετε προβλέψει κάποιο συγκεκριμένο προπολογισμό, μιλήσατε για συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσει, ε, ε, μιλήσατε για έρευνε, για μελέτε, ε, δημοσκοπήσεις. Έχετε κάποιο προπολογισμό που έχετε δεσμεύσει για μια τέτοια πρωτοβουλία. Κατά τα άλλα, σα ευχαριστώ. Ξέρετε, η τεχνολογία έχει προοδεύσει πολύ πιο γρήγορα από το ρυθμό διανομή των πληροφοριών στους πολίτες. Ευχαριστώ. ο ε, κύριος ε, Γκόκα, ε, μπορείτε να εξηγήσετε ποιος, σε ποιο βαθμό συνεργάζονται τα κράτη-μέλη μεταξύ τους αυτή τη στιγμή και πώς λειτουργεί αυτή η συνεργασία πρακτικά. Θεωρείτε ότι τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτή την οδηγία θα βοηθήσουν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Επίσης αναφέρατε ήδη ότι η σημερινή συζήτηση που γίνεται για αυτή την οδηγία θα αποδειχθεί ε, ουσιώδη για τις μελλοντικές εργασίες της ΕΝΗΣΑ. Θα γνωρίζετε πιθανώς ότι ε, αυτή η οδηγία εμπεριέχει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ΕΝΗΣΑ. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε στα μέλη της Επιτροπής αυτής εδώ πώς μπορεί να χρησιμεύσει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια των Δικτύων των Πληροφοριών, η ΕΝΗΣΑ, για θέματα ασφαλείας στα κράτη-μέλη και ειδικότερα για την αντιμετώπιση των ε, απειλών στον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Κάρλας. Ευχαριστώ. Μπορεί η ερώτησή μου να είναι ανόητη, αλλά εγώ θα την θέσω. Αναρωτιέμαι. Διάβασα τα, ε, τις εργασίες τα όσα κάνετε, αλλά δεν κατάλαβα για ποιον εργάζεστε. Ε, ποιο είναι το κοινό σας, ε, μπορείτε να το αναλύσετε λίγο. Και δεύτερον, από ό,τι κατάλαβα να πτήσετε κάποιες βασικές διαδικασίες που μπορούν να υιοθετήσουν και επιχειρήσεις. αφού έχουν έτσι τα πράγματα υιοθετούν τα κράτη και οι επιχειρήσεις στις βέλτιστες πρακτικές. Πριν από μερικές εβδομάδες ε, είχαμε μια εκδήλωση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπου μίλησαν διάφοροι εμπειρογνώμονες. Και αυτό που ανακαλύψαμε με πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο πιο αδύναμος κρίκος είναι ο άνθρωπος, ο χρήστης. Μιλήσατε λοιπόν για την εκπαίδευση, πιστεύω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, όσο και αν έχουν εξελιχθεί τα συστήματα από τεχνολογική άποψη, αν ο κόσμος ε, ε, εξακολουθεί να γράφει τους κωδικούς του πάνω σε ένα post-it, δεν χρησιμεύει εξέλιξη της τεχνολογίας. Και επίσης άλλη μια ερώτηση τώρα που σχετίζεται με όλα αυτά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τι κάνουν με τις βέλτιστες πρακτικές ε, στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε αυτά εδώ τα κτίρια γιατί ένας εμπειρογνωμόν είπε σε εκείνη την εκδήλωση ότι όταν μπαίνει σε αυτό εδώ το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σβήνει το Wi-Fi και δεν χρησιμοποιεί το έξυπνο τηλέφωνο του διότι υπάρχει κακόβλο λογισμικό παντού εδώ στο κτίριο αυτό και εμείς ε, φρίξαμε που το ακούσαμε. Οπότε το ερώτημά μου είναι πώς αντιμετωπίζουμε τα όλα πράγματα, όλη αυτή την κατάσταση εδώ. Έχει κανείς κάποια ερώτηση. Όχι, θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Δεν μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η απόψη σας για τη συνεργασία με άλλα μέρη του κόσμου στη στρατηγική για την ενέα ψηφιακή αγορά που συζητήσαμε με την Κομισιόν νωρίτερα. Ε, η Κομισιόν εστιάζεται στη βελτίωση των προτύπων πόσο σημαντικό θα ήταν να μην έχουμε μόνο ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά παγκόσμια για ζητήματα όπως το υπολογιστικό νέφος και η σχετική ασφάλεια ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια είναι τα ωφέλη αν αποφασίσουμε να διευρύνουμε την προσέγγιση πέραν της Ευρώπης ε, μέσω της συνεργασίας μπορείτε να μας πείτε την αψή σας πώς θα μπορούσε η ΕΝΗΣΑ και οι εμπειρογνώμονες της να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με άλλα μέρη του κόσμου ε, για να βρούμε πιθανά στομή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ξεκινώ με τον κύριο Σβάπ. Ρωτάτε για την ε, πλατφόρμα πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος. Δεν είμαι σίγουρος ότι πολλοί τη γνωρίζουν. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα. Δεύτερον, δεν έχουμε συγκεκριμένες διαδικασίες. Ε, κάποιες. Ε, ε, κάποιες έχουμε ελάχιστε, αλλά πολλές από αυτές λείπουν. Οπότε απαντώ και στην ερώτηση και για τον προπολογισμό ταυτόχρονα, γιατί έχει σχέση. Ε, οι δράσεις ευαισθητοποίησης. Στην ε, εντολή μας έχουμε 48 μονοθέσεις. Έχουμε ένα μόνο άτομο στο προσωπικό μας για την ευαισθητοποίηση από τις 48, 48 θέσεις. Ε, οπότε με τον προπολογισμό μας πληρώνουμε ε, τις ε, δαπάνες μετάβασης, αποστολών γενικά, ε, εκτύπωσης, φυλαδίων κλπ. Ε, υποστηρίζουμε δίκτυα στα κράτη-μέλη, μαζί με τα θεσμικά όργανα για την Κομισιόν βέβαια, και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και οι, οι, πρωτοβουλίες υποστηρίζονται οικονομικά και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι περισσότερες δραστηριότητε μπορώ να πω ότι παίρνουν χρηματοδότηση και από τις κυβερνήσεις αλλά κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε είναι μια καλή προσέγγιση ιδιωτικού δημόσιου τομέα, κοινή συνεργασία. Τώρα, στην Ενίσα θα χρειαζόμασταν περισσότερο προσωπικό για να κάνουμε κάτι παραπάνω. Η λογική είναι να έχουμε πολλαπλασιαστικό ε, αποτέλεσμα πάντως. Αναφερθήκατε και στην οδηγία ε, ασφάλειας των ε, δικτύων και των πληροφοριών. Την οδηγία NIS. Το είπα και πριν, η δύναμη της ΕΝΙΣΑ είναι να στηρίξει την εφαρμογή των οδηγιών της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, μιλώντας με τις κυβερνήσεις και με τον ιδιωτικό τομέα. Και όταν μιλάμε για ε, πρότυπα, ε, είναι Πολύ σημαντικό, σημαντική δράση μας. Αλλά, κοιτάξτε τον τομέα της τεχνολογίας προφορίας τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Νοτιοανατολική Ασία σε πολλούς τομείς. Αν θέλουμε να μπορούμε να επηρεάσουμε τα πρότυπα, θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά στα διεθνή όργανα προτυποποίησης. Κοιτάξτε την Nokia. Η Nokia πουλήθηκε στην Microsoft, το κινητό κομμάτι της. το κινητό κομμάτι της ε, Siemens εξαφανίστηκε, έκλεισε. Οπότε αυτές οι εταιρείες που, ήταν ευρωπαϊκές, που είναι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν συμμετέχουν και άρα δεν επηρεάζουν ε, τα πρότυπα που δημιουργούνται. Τα standards. Στην Ευρώπη έχουμε τη SEN, τη SENELEC και συνεργαζόμαστε μαζί τους. Οπότε ως ενίσα προσπαθούμε σε στρατηγικό επίπεδο να επηρεάσουμε τα πράγματα και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ε, η οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή που περάσαμε πέρσι και προσπαθούμε να δούμε με τη Elec ποια θα πρέπει να είναι τα πρότυπα, ποιες θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Οπότε σε ορισμένου τομεί μπορούμε να κάνουμε κάτι, σε άλλου όχι. Μετά, ερώτηση για την ανταλλαγή δεδομένων. Ξέρετε ότι αυτή είναι, αυτό είναι από τα βασικά προσκόμματα της οδηγίας NIS. Από πλευρά ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων, ε, τις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για εθνικό συμφέρον. Η ασφάλεια εξαρτάται εξαρτάται από το πώς τη βλέπουν τα κράτη-μέλη σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε φτάσει την οριμότητα που χρειάζεται για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε τέτοιου είδους ευαίσθητες πληροφορίες ε, σε κανονιστικό επίπεδο. Όλα λειτουργούν αυτή τη στιγμή ακόμα με βάση την εμπιστοσύνη και τις προσωπικές σχέσεις. Δεν έχουμε καταστήσει υποχρεωτική διανόμου αυτή την ανταλλαγή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και θέλω να το δούμε με δύο τρόπους. Έχουμε το αρθρο 33 13α που είναι ε, του, του πακέτου τηλεπικοινωνιών ε, που προβλέπει τις ε, ε παραβάσεων και ε, κάθε χρόνο δημοσιεύεται ένα έγγραφο. Ε, έχουμε συζητήσει με τα Υπουργεία ποιες είναι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται και ποια είναι η πραγματικότητα. Εσείς ψηφίσατε ένα κανονισμό και ε, τις λεπτομέρειες αφήσατε να αποφασιστούν στο φάση της ε, εφαρμογής. Και τι έγινε τελικά, οι πληροφορίες που ανταλλάσσουν είναι ελάχιστες πια. Για όλη την Ευρώπη α, ενημερωνόμαστε για 100-120 περιστατικά το χρόνο μόνο, τίποτα άλλο. Γιατί δεν ανακοινώνονται τα πάντα. Γιατί πολύ συχνά οι επιχειρήσει και οι κυβερνήσει δεν θέλουν να τα ανακοινώνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τα δημοσιοποιούν. Οπότε το θέμα είναι τι θα κάνουμε και με αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε κάθε κυβέρνηση να πάρει ε, τις αποφάσεις της. Η Κομισιόν θα αξιολογήσει το πακέτο επικοινωνιών σύντομα, αλλά αν δούμε το θέμα από το ευρωπαϊκό επίπεδο, βλέπουμε ότι το κάθε κράτος μέλος λέει αυτό την δική μου χώρα, εγώ βλέπω με το δικό μου τρόπο την ασφάλεια, οπότε αρνούνται να ανταλλάξουν ε, πληροφορίες. Ε, προστασία δεδομένων. Υπήρχε και γι' αυτό μια ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και συνδυάζω αυτό το ερώτημα με το ερώτημα από τη Ρουμανίδα συνάδελφο. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είστε 18χρονος και παίρνετε δίπλωμα οδήγηση και οδηγείτε με χίλια. Οπότε ε, ένα θέμα είναι να δώσουμε την άδεια οδήγηση και ένα άλλο να μάθουμε σε κάποιον, άνθρωπο νέο πώς ε, να λειτουργήσει και να οδηγεί στο αυτοκίνητο. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και συστήματα ασφάλειας όπως η ασφάλιση του αυτοκινήτου, έχουμε κυρώσεις, έχουμε ελέγχους που αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης αν κάποιος οδηγεί γρήγορα κλπ. Αυτό δεν ισχύει για τα συστήματα πληροφοριών. Ε, εγώ όταν ήμουν μικρός ερχόντουσαν αστυνομικοί στα σχολεία και μου λέγανε πώς να οδηγώ το ποδήλατό μου. Οπότε υπάρχουν οι προκλήσεις, αλλά δεν ετοιμάζουμε τους ανθρώπους να τις αντιμετωπίσουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και ακόμα και όταν το κάνουμε <clears throat> γίνεται κατακαιρματισμένα σε τοπικό επίπεδο κλπ. κλπ. Ε, αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση αυτή, η επιμόρφωση αυτή δεν προβλέπεται υποχρεωτικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και πολλοί συναγωνείς δεν μπορούν να την προσφέρουν. Μετά, θα πρέπει να ενημερωθούν και οι κυβερνήσει, ασφαλώ. Ο δικό μου δισταγμό είναι ότι ε, σε πολλές περιπτώσεις ενημερώνουμε το κοινό και ενημερώνουμε και τις κυβερνήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το αντίστοιχο θέμα θα είναι προτεραιότητα για αυτούς, για τους πολιτικούς. Καμιά φορά είναι, αλλά συνήθως η ασφάλεια των δικτύων δεν είναι πολιτική προτεραιότητα. Οπότε όσο και να τους ενημερώσουμε τι θα γίνει. Μετά, συνεργασία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά με μικρου βελληνικούς πρωτοβουλίες. Ξέρω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που ε, χρησιμοποιούν συστήματα αλληλοδιδασκαλίας. Είναι καλές πρακτικές, οι οποίες ανταλλάσσουμε, προσπαθούμε να τις διευρύνουμε. Προσπαθούμε να μεταφράσουμε από τη μια γλώσσα στην άλλη αυτές τις εμπειρίες. Επίσης με ερώτηση κυρία Κάλλας για ποιον δουλεύουμε. Είναι θεμητή ερώτηση. Νομίζω ότι αναφέρθηκα σε αυτό λίγο στην αρχή. Είπα ότι στις κυβερνήσεις έχουμε πολύ καλή δομή, που ξέρουμε ποιον θα μιλήσουμε, με τη, στο, στον ιδιωτικό τομέα λίγο λιγότερο. Οι βασικοί μας πελάτες εκεί είναι η υπεύθυνοι ασφαλεία των επιχειρήσεων. Έχουμε ένα-δύο παραδείγματα. Ε, ε, στο, στην υπολογιστική νέφους, για παράδειγμα, έχουμε εκδώσει πολλές συστάσεις, έχουμε προτείνει ένα σύστημα πιστοποίησης, ε, υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες εφάρμοσαν αυτές τις συστάσεις και έχουμε μάλιστα και ε, Έχουμε και έναν, δύο ε, παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους, υπολογιστικού νέφους που έχουν αυτοπιστοποιηθεί με βάση αυτές τις διαδικασίες. Οπότε για ορισμένα πράγματα έχουμε δίκτυα από παλιά, ανταλλάσσουμε πληροφορίες κλπ. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει και δίκτυα όπως αυτό των ε, αξιωματούχων ε, άμεσης αντίδρασης σε ε, εκτακτές περιστάσεις. Υπάρχει ένα σε κάθε κράτος μέλος. Οπότε ε, προσπαθούμε να δικτυωθούμε και να δικτυώσουμε. οπότε η ασφάλεια θα πρέπει να εξασφαλίζεται καταρχήν όσο πιο κοντά γίνεται στους κινδύνους. Κοιτάξτε την Europol. Η Europol, μάλλον ε, οι εγκληματίες συλλαμβάνονται στην πόλη στην οποία ζουν, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται και διεθνή συνεργασία. Οπότε το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην περίπτωση της ασφάλειας των δικτύων. Η κάθε χώρα, η κάθε οργάνωση κλπ. θα πρέπει να έχει το δικό τη ε, ε, δίκτυο ασφαλεία, το δικό τη σύστημα ασφαλεία, αλλά ταυτόχρονα να συνεργαζόμαστε και σε διεθνέ επίπεδο. Οπότε τα κράτη-μέλη και ο ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να είναι οι πρώτοι παίκτε και εμείς να τους βοηθάμε. Ε, έχουμε δει επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις και εναντίον του τομέα των μέσων ενημέρωση των media. Απ' την άλλη μεριά δεν είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς. Εμείς στην ΕΝΙΣΑ ε, συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, εταιρείε ε, που παράγουν προϊόντα σχετικά με την εξασφάλιση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών. Και αυτές οι εταιρείε έχουν πελάτες. Λοιπόν, φτάνοντας εμείς σε αυτές τις εταιρείε και ενημερώνοντάς τις, αυτές μπορούν να ενημερώσουν τους πελάτες τους. Οπότε αυτό έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, αλλά και αυτό παίρνει χρόνο. Έχουμε επίσης δίκτυο αξιωματούχων ε, ασφάλειας τεχνολογίας των πληροφοριών με τα κράτη-μέλη και με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελειώνω. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το υπολογιστικό νέφος. Ε, τα smartphones και τα κινητά τηλέφωνα δεν χρονολογούνται από πολύ παλιά. Είναι κάτι σχετικά καινούριο. Και τι βλέπουμε. Οι μεγάλοι παίκτες στις ΗΠΑ κοινωνική δικτύωση, ε, μηχανές αναζήτησης κλπ. Ε, υπήρχαν από πιο παλιά, αλλά και πάλι όχι πολύ παλιά, οι Κινέζοι τα τελευταία 10 χρόνια, μπαμπά κλπ. Εμείς το έχουμε χάσει αυτό στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Η ITU είναι μια παγκόσμια οργάνωση. Είναι η Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Εκεί δεν επηρεάζουμε πολύ τα πράγματα, δυστυχώ. Πια. Οπότε, ως Ευρώπη, πού μπορούμε να επηρεάσουμε. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό και, και εσείς ως Επιτροπή να δείτε το μέλλον του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της ε, ε, τεχνολογίας των πληροφοριών και πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλει κανείς να κάνει δεύτερη ερώτηση. Χρόνο έχουμε. Έχουμε τον κύριο Λάμπερτς, τον κύριο Φανίστηλ Ρόι. Ναι, ευρύτατο θέμα. Με προβληματίζει η τοποθέτηση ότι μπορεί να χάσαμε μερικούς αγώνες, αλλά ίσως όχι τον πόλεμο. Πού βλέπετε εσείς τα πλεονεκτήματα στη δυτική χώρα των κάτω χωρών. Έχουμε πολύ μεγάλο δυναμικό. Και πρέπει για να εξασφαλίσουμε την κυβερνοασφάλεια να έχουμε προσωπικό ικανό, όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και να είναι αρκετά ισχυρός να πιάνει τον κλέφτη. Μιλήσατε για ένα σύστημα κατάρτισης, επιμόρφωσης και ξέρουμε ότι έχουν γίνει πολλές εβδομάδες για το coding ώστε εγκαίρως τα παιδιά και στην πρωτοβάθμια και ε, εκπαίδευση ήδη να εξοικειωθούν με την ε, ανάπτυξη κωδικών. Πού μπορεί να φτάσει αυτό, πόσο μπορεί να ενσωματωθεί στην πραγματική εκπαίδευση και ως προς τις προσλήψεις. Εάν χάσετε από το ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί να μην χάνετε μόνο σε επιχειρησιακό επίπεδο. Χάνετε διπλά. Χάνουμε διπλά καλύτερα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Παρακαλώ από την DigiConnect, Connect ο κύριος Μπριν Κάταν έχει κάτι να μας πει. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. όπως είπατε, και εμείς παρακολουθούμε τις συνεχιζόμενες συζητήσεις για την οδηγία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Και περιμένουμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ελπίζουμε ότι θα στεφθεί με επιτυχία η διαπραγμάτευση της οδηγίας, ώστε αυτή να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών το ταχύτερο δυνατό. Για το υποσυζήτηση θέμα, οδηγία για, την οικουμενική υπηρεσία και ιδιαίτερα το ζήτημα της πλατφόρμας και της προσφοράς πληροφοριών στον πολίτη εν γέννη. Πρόκειται πιστεύω για ένα εργαλείο το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου. Για μας, δυστυχώς, ως Επιτροπή, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο δράσης. Νομικά τουλάχιστον δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, να παρέμβουμε. Τι κάνει όμως η οδηγία. Η οδηγία δίνει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη, την εξουσία καλύτερα, να καλέσει όλους τους παρόχους πληροφοριών που εμπλέκονται στις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες. Όλες τις ε, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών δηλαδή, όλες τις επιχειρήσεις που καλύπτουν τον τομέα. Μπορεί να τις ε, καλέσει λοιπόν να προσφέρουν πληροφορία ως ε, τμήμα οικουμενικής υπηρεσίας όλες τους πελάτες. Και το ίδιο θα το δείτε στα κομμάτια που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια. Είναι όντως πολύ δαπανηρή η πρόσβαση στην πληροφορία. Ταυτόχρονα όμω πρόκειται στην ασφάλεια τη πληροφορία, αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για ένα εργαλείο υπαρκτό, ένα εργαλείο που προβλέπει οδηγία, ένα εργαλείο το οποίο δυστυχώ δεν αξιοποιείται επαρκώς, ενώ δεν κοστίζει σε εμά και τα κράτη-μέλη τίποτα, διότι υφίσταται η υποχρέωση για τον πάροχο με τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει να προσφέρει τις πληροφορίες αυτές στους πολίτες. Άρα, καταρχήν μπορώ να πω ότι δεν γνωρίζουμε να υπάρχει κρατός μέλος το οποίο να υλοποιεί αυτήν την διάταξη της οδηγίας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Και επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης. Πρέπει να έχουμε όμως υπόψη ότι αναμένεται η αναθεώρηση της οδηγίας για τις ε, ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες. Γι' αυτό δεν θέλουμε και να προδικάσουμε τίποτα μπορεί να προκύψει από τις συνομιλίες αυτές. Προς το παρόν έχουν υποχρέωση μόνο τα κράτη-μέλη ως προς το εξή, εάν θέλουν, μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο. Αυτή είναι η υποχρέωσή τους. Και από ό,τι γνωρίζουμε εμεί τουλάχιστον δεν έχουν αξιοποιήσει τη διάταξη αυτά τα κράτη-μέλη. Το μέσο όμως αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να ενημερώνεται ο πολίτη για τα κύρια ζητήματα της ε, προστασίας του ειδικού βίου, της ασφάλειας, γενικά ω μέσο ευαισθητοποίηση. Η Πρόεδρος. Θέλετε να επανέλθετε. Κάποιος άλλος συνάδελφο θέλει να κάνει σχόλιο. Αν μου επιτρέπετε, θέλω κι εγώ να πω ότι υπάρχουν πολλές επιτυχημένες νέες επιχειρήσεις. Στη Φιντέκε παραδείγματι στην πατρίδα μου έχουμε ιδιαίτερες επιτυχίες. Η Γκεμάλτο η οποία κάνει και είναι παγκοσμίου εμβελίας ε, επιχείρηση, μικροτσίπ, ε, Άρα υπάρχουν τομεί στου οποίου οι Ευρωπαίοι έχουν την πρωτοκαθεδρία. Α το θυμόμαστε αυτό για να υποστηρίζουμε και τι θετικέ πτυχέ, όχι μόνο τα αρνητικά. Κύριο Χέρμπερτ, δεν θα διαφωνήσω με αυτό που είπατε. Αλλά δεν θέλω να το ονομάσω αυτό που λέω σήμα αφύπνισης δεν αλλάζει τίποτα με το να έχουμε μια-δύο καινούριε επιχειρήσει. ή ούτε καν με το να μην έχουμε το κατάλληλο σύνολο δεξιοτήτων. Γιατί παραδείγματι έχουμε πολλού Ρουμάνους στο προσωπικό μας ύψη τη ε, κατάρτισης, ε, κανούς μπορούν να αξιολογήσουν και να κάνουν πολύ καλή δουλειά με την ΕΝΙΣΑ. Αυτό που έχω να πω λοιπόν είναι ότι πρέπει να εστιαστούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι βλέπουμε τη διαφορά με τι Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαφορά ποια είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν 300 εκατομμύρια πολίτε με ένα νόμισμα και τη μέρα που θα ξεκινήσει μια startup στο Texas, στο Silicon Valley, θα αρχίσει να λειτουργεί το application που θα παραγάγει αύριο αμέσω σε όλο τον κόσμο, στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Αυτή είναι η κρίσιμη μάζα. Στην Ευρώπη έχουμε 28 διαφορετικά κράτη-μέλη, 18 λέει ο στην Ευρωζώνη, έχουμε τον web servers στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία που μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση αλλά να ξεκινήσει εκεί δεν μπορεί να απολύσει ε, το startup της στην ε, Πορτογαλία ή στην Πολωνία. Αλλιώς θα χρειάζεται να κάνει μια σειρά από διαφορετικές διαδικασίες για το κάθε κράτος μέλος. Και βέβαια η κρίσιμη μάζα αλλοιώνεται και όταν μεγαλώνει αυτή η επιχείρηση άλλο είναι τα 10, 20, 30 εκατομμύρια για startup. Αν κάποιο χρειάζεται 100, 200 εκατομμύρια για να ξεκινήσει μια δουλειά, αυτό στην Ευρώπη είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί. Φιλανδικέ ή γερμανικέ επιχειρήσει που να το έχουν ε, σαν δυνατότητα, τότε αμέσω εξαγοράζονται από αμερικανικέ. Και αν σα ενδιαφέρει, σα στείλω πιο λεπτομερή στοιχεία για το τι συμβαίνει. Άρα το ζήτημα δεν είναι η εκπαίδευση και το know-how, η τεχνογνωσία. Τα έχουμε αυτά όλα. Έχουμε πάρα πολύ καλέ επιδόσει. Η ανάπτυξη όμω δεν ε, μένει στα χέρια των Ευρωπαίων. Δεν θα αγοράσουν αυτές τις νέες επιχειρήσεις Ευρωπαίοι. Αλλά οι Αμερικανοί που έχουν την κρίσιμη μάσα. Γι' αυτό σα λέω, κοιτάξτε τι γίνεται στι ΗΠΑ, κοιτάξτε τι γίνεται στην Κίνα που μπορεί να έχουν διαφορετικά κοινωνικά συστήματα, αλλά έχουν πολύ ανάλογη ανάπτυξη στον χώρο τη τεχνολογία. Έχουμε λοιπόν το δυναμικό, αλλά δεν έχουμε την ανάπτυξη. Και το κρίσιμο ζήτημα είναι τώρα, από εδώ και μπρο στο μέλλον, που θα εξαρτώνται τα πάντα από την τεχνολογία την ψηφιακή, και θα χρειάζεται να αγοράζουμε τα πάντα από ολίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Ερωτηματικό. Ευχαριστώ πολύ και που μας υπενθυμίσετε ότι χρειάζεται μια πραγματική ενιαία αγορά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Ασφαλώς θα υπάρξουν και δεμερείς συνομιλίες. Ε, ευκαιρία στο θύσεις. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Και έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση και σε σχέση με τον κίνδυνο στη Λυπή Ευρώπη. Στο ταχύτερο δυνατό ξεκινούμε συνεδρίες των συντονιστών, εκτός και αν έχετε έτερον για τα διάφορα. Όχι. Σας ευχαριστώ θερμά.